Χρόνια σας πολλά. Η Εστονία γιορτάζει την εκατοστή της επέτειος στις 24 Φεβρουαρίου του 2018 και η χώρα σας ε, σκοπεύει να ε, ε, έχει ένα θεματολόγιο με θέμα ενότητα μέσω της ισορροπίας, unity through balance, το οποίο θα γεφυρώσει τους τομείς οικονομίας, της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας. Σας ευχόμαστε καλή τύχη για την πρώτη σας προεδρία, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της ήδη από το 2012. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν θα θέλαμε κύριε Σβέν Μίξερ να μας πείτε τους βασικούς στόχους σας για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Φαντάζομαι ότι θα επικεντρωθείτε στη διεύρυνση, στην Τουρκία, τη Μεσόγειο. Ε, ίσως θα θέλετε να μας πείτε και κάτι για τη σύνοδο του Ιστεργέστης, η οποία θα γίνει αύριο, ξεκινάει μάλλον αύριο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσεγγίσουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προτείνω λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό και μετά θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό το αργότερο στις 4, γιατί από εκεί και πέρα περιμένουμε τη Χέλγα Σμιτ για να μας ε, πει κάποια πράγματα πριν από το FAC. Ε, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστερ αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Εκτιμώ ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας για τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας ε, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ε, και της διεύρυνσης, ε, πολλό δε μάλλον διότι πριν από δύο μοίρες είχαμε τουλάχιστον 10 από τους 15 υπουργούς της Εστονίας εδώ στις Βρυξέλλες, οι οποίοι ήρθαν και μίλησαν στις διάφορες επιτροπές για τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Ε, Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες εναλλακτικέ λύσεις αντί να έρθετε να ακούσετε εμένα σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και ε, χαρά να είμαι εδώ να συζητώ μαζί σας για τα θέματα αυτά. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις πολύ καλές επαφές που έχουμε ήδη ε, συνάψει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά εκτιμώ και την ε, αγαστή συνεργασία ιδίως με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Πρόεδρε, συναντηθήκαμε το Μάρτιο και νομίζω ότι αυτή η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι καταφέραμε να καταρτήσουμε το θεματολόγιο για την Προεδρία και μου έδωσε και μια πολύ καλή αντίληψη των προσδοκιών ε, των δικών σας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γέννη για την Προεδρία. Ε, βεβαίως ε, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα καθημερινά και θέλουμε να είμαστε και αρκετά ευέλικτοι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, όλες τις σχετικές εξελίξεις ε, ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στην γειτονία της Ευρώπης και νότια και ανατολικά. Επίσης, θα ήθελα να σε χαρώ τη Μαλτέζικη Προεδρία για την εξαιρετική της δουλειά. Το προηγούμενο εξάμεινο είχαμε εξαιρετική συνεργασία, εξαιρετικές επαφές με τους Μαλτέζους συναδέλφους και φυσικά ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες ε, με τους ε, εταίρους μας, το τρίο, τη Βουλγαρία και την Αυστρία δηλαδή. Την Άνοιξη η Εστονία θα κλείσει 13 χρόνια από τότε που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να πέρασε αυτός ο χρόνος, αλλά αν εξετάσω τι κάναμε πριν την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τη χώρα μας ε, για την ένταξη ε, και να πληρούμε όλα τα κριτήρια. Ε, κοιτώντας βέβαια πίσω μπορώ να πω ότι και η χώρα μας και οι πολίτες φυσικά της χώρας ε, εποφελήθηκαν ε, των οικονομικών ευκαιριών και φυσικά και της σταθερότητας που προέρχεται ακριβώς από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, το 1997 ή μόλις γιορτάσαμε και την 60η επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης ότι έχαμε έξι δεκαετίες ε, ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας χωρίς προηγούμενο και η χώρα μου κατάφερε να συμμετέχει τα τελευταία 13 χρόνια σε αυτό το όραμα. Ε, Πέρσι όμως, ε, μετά από την ψηφοφορία για το Brexit, ε, έγινε σαφές ε, για όλους ότι αυτή η αισιοδοξία και αυτή η θετική αίσθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι κοινό σε όλους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρχίζουν να ρωτούν αρκετές ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς αυτοί οι φόβοι οι οποίοι οξύνθηκαν μετά από το Brexit ε, κατάφεραν σιγά σιγά να υποχωρήσουν και σήμερα υπάρχει λίγο περισσότερος ενθουσιασμός ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι είχαμε προηγουμένως ε, πριν από ένα χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό αντανακλάται και στους θετικούς συσχετισμούς που έχουμε στην οικονομία μας. Υπάρχει ανάκαμψη και πάλι. Ε, αισιόδοξο τρόπο ε, να βλέπουμε τα πράγματα που διαφάνηκε και μετά από τα πρόσφατα αποτελέσματα στις εκλογές. Ε, βέβαια δεν έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, ζούμε σε χαλεπούς ε, καιρούς, ε, απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν και φυσικά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, το σύνθημα της Εστονικής ε, Προεδρίας είναι ενότητα μέσω της ισορροπίας, unity through balance. Ε, πρόκειται για πολύ μεγάλη υποστήριξη για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Έννοιας και του Ευρωπαϊκού Οράματος, καθώς επίσης και σεβασμός της διαφορετικότητας, ο οποίος θεωρώ ότι αποτελεί αυταξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και Υπάρχει πληθώρα συμφερόντων και ενδιαφερόντων ε, και διαφορετικές προτεραιότητες ε, όταν ε, συζητούμε για 28 κράτη-μέλη τα οποία σύντομα θα γίνουν 27. Πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε τη δέουσα ισορροπία μεταξύ των ατομικών και μεμονωμένων συμφερόντων ορισμένες φορές των κρατών μελών της Ένωσης και του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συνεχίσει η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προχωρήσουμε και γι' αυτό και έχουμε καταλήξει σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες, τις οποίες έχουμε δομήσει το θεματολόγιό μας. Καταρχάς, μια ανοιχτή και καινοτόμα ευρωπαϊκή οικονομία, ε, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών και των κοινωνιών. Δεύτερον, μια ασφαλή και σίγουρη Ευρώπη. Ε, πιστεύουμε στην έννοια ε, της ε, ασφάλειας και θεωρούμε ότι είναι αδιαίρετη και οι εξωτερικές και οι εσωτερικές πτυχές της ασφάλειας αλλά και είναι και αδιέρετη και ε, με τη γεωγραφική της έννοια, διότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, εξελίξεις οι οποίες ε, εκτιλήσονται πολύ μακριά από εμά μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές επιπτώσεις και επιρροή για την ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσους και προφανείς τρόπους. Τρίτον, κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως εστονό, μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι το ψηφιακό θεματολόγιο, Πρόκειται για ένα ευρύ θέμα που καλύπτει θέματα όπως ε, την ψηφιακή οικονομία και την ελεύθερη ε, ροή πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια και ούτω καθεξής. Και βεβαίως μια Ευρώπη βιώσιμη που περιλαμβάνει τους πάντες. Αυτή είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα και ο Πρωθυπουργό μας ε, παρουσίασε το θεματολόγιο την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Θέλουμε να προωθήσουμε ε, το θεματολόγιο αυτό συνολικά στη διάρκεια του εξαμήνου ε, και να καταλήξουμε σε συνένεση όπου υπάρχει και όπου δεν υπάρχει να δούμε τι θετικές ε, εξελίξεις μπορούμε να έχουμε για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και το θεματολόγιο μας εκεί, θα ξεκινήσω με τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι στο επίκεντρο του θεματολογίου μας διότι πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μοχλούς μεταρρυθμίσεων στις χώρες οι οποίες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να γίνουν μια μέρα μέλη της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στην ελευθερία, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου και επομένως περιμένουμε ε, οι αξίες αυτές να είναι κοινέ ε, για όλες τις υποψήφιες χώρες. Αλλά φυσικά ε, δεσμευόμαστε στην εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης η οποία θα βασίζεται στις ε, ε, συγκεκριμένες αρχές και στις αξίες και στους όρους που υπάρχουν. Επισκέφθηκα κάποιες χώρες στους τελευταίους μήνες, ξεκίνησα με τα Δυτικά Βαλκάνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συζητήσει βεβαίω την κατάσταση των Δυτικών Βαλκανίων επανειλημμένω. Το Μάρτιο τα κράτη-μέλη ε, επιβεβαίωσαν σαφώ την ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες της περιοχής. Ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επεσήμασαν τη σημασία των μεταρρυθμίσεων, των καλών σχέσεων και ε, τη περιφερειακή συνεργασία. Όλα αυτά είναι απόσπαστα στοιχεία τη διαδικασία ολοκλήρωση και φυσικά και τη διαδικασία σταθεροποίηση. Και πρέπει εδώ να αναφέρω ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι διαπραγματεύσεις με όλες τις υποψήφιες χώρες ε, πόρο απέχουν από την ολοκλήρωση, αλλά ε, έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ε, και τα καταγράψαμε αυτά και στη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας, διότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσαμε να ανοίξουμε και σε κάποιες περιπτώσεις να κλείσουμε προσωρινά κάποια κεφάλαια για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις και προφανώς ελπίζουμε και να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε επιπλέον κεφάλαια στη διάρκεια της δικής μας της Προεδρίας. Οι πιο σημαντικοί τομείς στους οποίους πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η πρόληψη της διαφθοράς, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, και ε, ταυτόχρονα αναμένοντας αυτά τα αποτελέσματα από τις υποψήφιες χώρες πρέπει να είμαστε και βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή θα πληρούνται οι προϋποθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να κάνει αυτό που της αναλογεί δηλαδή ε, να καλύψουμε και εμείς τις δικές μας τις υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή οι χώρες ε, ε υποψήφιες έχουν κάνει αυτά που ε, πρέπει. Μόνο έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση. Δύο λόγια τώρα για την κάθε χώρα της περιοχής. Το Μαυροβούνιο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ε, ε, διαπραγματεύσεων προσβλέπουμε στην πρόθεση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στη διάρκεια της Προεδρή αλλά θέλουμε να παρακολουθήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει το Μαυροβούνιο στον τομέα του κράτους δικαίου. Θέλουμε επίσης να έχουμε μια σταθερή πολιτική διαδικασία. Ε, θα όλα τα πολιτικά κόμματα να επιστρέψουν στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, στο Κοινοβούλιο, προκειμένου η πολιτική συζήτηση να επιστρέψει στα θεσμικά όργανα, εκεί που ανήκει και όχι να ποικοτάρουν αυτά τα όργανα ε, και να διαδηλώνουν στους δρόμους. Ε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο έγινε μέλος του ΝΑΤΟ ε, πρόκειται για μια διαδικασία που προσπάθησαν ε, να ε, πυρπολίσουν κάποιοι ακόμα και το περασμένο φθινόπωρο και να εκτροχιαστεί όλη η διαδικασία αλλά καταφέραμε τελικά να ολοκληρώσουμε επιτυχώς αυτή τη διαδικασία και αυτό προσδίδει αξιοπιστία στην πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Σερβία τώρα νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ο νέος Σέρβος Πρωθυπουργός πρέπει να ε, εντατικοποιήσει τις προσπάθειες. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος Βελιγραδίου-Πρίστινας και πρέπει να προχωρήσουμε όλες τις συμφωνίες οι οποίες έχουν επιτευχθεί, ήδη μεταξύ των διαφόρων πολιτικών κομμάτων όσον αφορά ε, τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις εκλογές στη χώρα. Δεν είναι πολύ εύκολα αυτά πάντα, αλλά πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους εταίρους μας ε, όλα αυτά τα στοιχεία. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς ε, στην επίσκεψή μου στη Σερβία, ο πρόεδρος μου υπενθύμησε ότι η διεύρυνση και η ένταξη της Σερβίας είναι ο, ο μόνος δρόμος για αυτούς ένα από τα κρίσιμα κεφάλαια φυσικά είναι το κράτος δικαίου. Και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ερβικές αρχές βεβαίως να προωθήσουν τα στοιχεία αυτά. Και όπως είπα και η εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό και ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με όλα τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βεβαίως και το Κοινοβούλιο. Και το Κοινοβούλιο υπήρξε πολύ δραστήριο και προωθεί τις μεταρρυθμίσεις ε, στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων για να μπορέσουν να συνεργαστούν όλοι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για το κοσφοπέδιο σας είπα ήδη ότι υπάρχει ο διάλογος Βελιγραδίου Πρίστινας οι πρόσφατες εκλογές ε, στο Κοσφοπέδιο δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά ελπίζω ότι ε, θα ε, γίνει σίγουρα και θα μπορέσει να προχωρήσει η νέα κυβέρνηση με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τον ευρωπαϊκό δρόμο και ενθαρρύνουμε το κοσυφοπαίδιο να εκμεταλλευτεί ε, αυτές τις δυνατότητες χρειάζονται προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς επίσης και στην εξομάλυνση των σχέσεων με τους γείτονες όχι μόνο με τη Σερβία αλλά και τη συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο η οποία είναι ακόμα εν αναμονή κύρωσης. Για την ε, Πογουδμού. Καλώς ορίζουμε τις εξελίξεις στην χώρα αυτή όπου επιτέλους που ορκίστηκε νέα κυβέρνηση μετά από πολύ χρόνο που χάθηκε και η κυβέρνηση υποσχέθηκε να ξαναξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις που είχαν καθυστερήσει και να εφαρμοστεί επίσης και η συμφωνία που υπεγράφει. Υπάρχουν ήδη κάποια ενθαρρύνματα ε, σημεία την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση έκανε ένα σχέδιο δράσης για τις μεταρρυθμίσεις αλλά σημαντικό είναι να προχωρήσει και η πολιτική διαδικασία και αναμένουμε να δούμε μια επικοδομητική διάθεση της ε, κυβέρνησης απέναντι στην αντιπολίτευση. Και προφανώς αναμένουμε οι αρχές να στηρίξουν το έργο του ειδικού εισαγγελέα. Επίσης, αναμένουμε να ενθαρρύνουμε την πρόοδο σε σχέση με το όνομα που καθυστερεί την ε, διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την διαδικασία ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ε, δηλώσεις από την νέα κυβέρνηση. Για την Αλβανία έγιναν οι εκλογές, ε, οι βουλευτικές ε, τον Ιούνιο και ελπίζουμε να υπάρξουν αποτελέσματα. Σημειώσαμε επίσης την σύσταση υπό όρους της Κομισιόν πέρσι για να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Προφανώς βεβαίω θα εξαρτηθεί από την πρόταση της ε, Κομισιόν και θέλουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον. Για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη προφανώς υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, να ενταθούν οι προσπάθειες για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αναμένουμε η χώρα να παραμείνει εντός της ε, διαδικασίας ε, και θα βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρουσία της αλλά η κύρια ευθύνη για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία βεβαίως είναι των αρχών και η διχαστική ρητορία που είχαμε δει στο παρελθόν δεν βοηθάει τη χώρα ούτε τον λαό ούτε την ευρωπαϊκή ένταξη. Η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα και σημαντικός εταίρος Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την επαφή και έναν ανοιχτό διάλογο με τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα πρέπει να παραμείνει νομίζω σε μια κατεύθυνση που θα στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και ανεξαρτήτως του τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πρέπει να παραμείνουμε αταλαντευτοί. Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια η συνεδρίαση στις 25 Μαΐου μεταξύ των Προέδρων Τούσκ, ε, Γιούνκερ και Τεγέννη και του Πρόεδρου Ερντοκάν μας έδωσε μια ευκαιρία να προχωρήσει ο διάλογος με τρόπο θετικό και όχι με αντιπαραθέσεις. Θέλουμε να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία στην αντιδρομοκρατία, ενέργεια, οικονομία και μετανάστευση και η δήλωση, η εφαρμογή της δήλωσης είναι κάτι το θετικό. Ήδη έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα συγκεκριμένα μειώθηκαν οι θάνατοι στη Μεσόγειο. Τότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και αν η Τουρκία θέλει να προχωρήσει στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αυτές είναι οι αξίες που θα πρέπει να σεβαστούν οι αρχές, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος ε, σχεδόν ο μισός πληθυσμός ψήφισε κατά των προτινόμενων αλλαγών. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην απογοητεύσουμε το κομμάτι αυτό των Τούρκων πολιτών. Όσον αφορά τώρα βεβαίως τις συνομιλίες για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Να, πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να δούμε τις ε, θετικές πτυχές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει όλες τις προσπάθειες και αναμένει από την Τουρκία να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο. Τέλος, για κάποια ζητήματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση με την πολιτική διεύρυνση. Πρώτα απ' όλα η μετανάστευση. Το θέμα αυτό απαιτεί μια συνολική προσέγγιση. Πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών, αλλά χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση να βρεθεί μια μόνιμη λύση στην μεταναστευτική κρίση. Είναι προτεραιότητα της Προεδρίας μας και νομίζω είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη υπουργική διάσκεψη στο Ταλίν την προηγούμενη εβδομάδα των Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συναντήθηκαν το θέμα της μετανάστευσης ε, στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, δηλαδή από τη Λιβύη στην Ιταλία, ήταν ε, πρώτο στην ημερήσια διάταξη και προφανώς θα παραμείνει το θέμα στο εξωτερικό μέτωπο προφανώς πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να αυξηθεί η αντοχή των κοινωνιών και των κρατικών δομών, των κοινωνιών εκείνων από που προέρχονται οι δομές αυτές. Την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνησή μας αποφάσισε να δώσει άλλο ένα εκατομμύριο από τον προπολογισμό της στο Ταμείο για την Αφρική. Προφανώς θέλουμε να εργαστούμε σκληρά για να προωθήσουμε τις δυνατότητες των σχετικών κρατικών νομών και τις ικανότητες των αφρικανικών χωρών να ελέγξουν τα σύνορά τους. Και βεβαίω εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να επεκτείνουμε τις δυνατότητες ε, των ε, επιχειρήσεων που προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και προφανώς θέλουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ε, αντιμετώπισης των πρακτικών πτύχων, καταγραφής και συνεργασίες με τους μετανάστες που κατευθύνονται προς τις ευρωπαϊκές ακτές και Βεβαίω η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό. Τέλος, για την ανατολική γειτονία. Και αυτή είναι μια προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Θεωρούμε ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην στήριξη της ε, μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στις έξι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να εδραιώσουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει. Έχουμε τις ε, συμφωνίες σύνδεσης ε, με τρεις από τις έξι χώρες και τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και οι πολίτες των τριών χωρών μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην Ευρώπη Τώρα, για τα υπόλοιπα έχουμε καταλήξει κάποιοι... Έχουν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες με την Αρμενία για μια νέα συμφωνία πλαίσιο και είμαστε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας νέας συμφωνίας με το Αζερβαϊτζάν. Ε, προφανώς για τη Λευκορωσία πρέπει να παρακολουθούμε τις εσωτερικές εξελίξεις, αλλά είδαμε πέρσι κάποιες ε, θετικές εξελίξεις, κάποια πιστοχώρηση φέτος αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε και την Λευκορωσία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ε, τώρα δεν θα ήθελα να επιμείνω στις σχέσεις μας με την Ρωσία και τις ε, διατλαντικές σχέσεις και κάποιες άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλεία της Ευρώπης. Ευχαρίστω να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα στην απάντηση στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε, Sven Mixer, για τις ε, ερωτήσεις της Τονικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Ε, θα κατέχει την Προεδρία του Συμβούλιου. Έχουμε 26 λεπτά στη διάθεσή μας για ανταλλαγή απόψεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ομιλητέ στον κατάλογο. Και Πρέντα, Μαυρίδες, Σελαμόν, Ζόφκο. Έχω 8 συναδέλφους και θα κλείσω τον κατάλογο. Δύο λεπτά ο καθένας και έχουμε 10 λεπτά για να απαντήσει ο υπουργό. Ο πρώτος, ομιλητή είναι φυσικά ο εσθονό συνάδελφο Τόνι Κίλεν. Ευχαριστώ πολύ. Με έχουν ενθαρρύνει πάρα πολύ οι προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας σχετικά με τη διεύρυνση, την ανατολική σχέση, την μετανάστευση και τα Δίκτυα Βαλκάνια. Αλλά όπως γνωρίζουμε, τελικά το αδιέξοδο εδώ, στη διαδικασία διεύρυνσης στα Δίκτυα Βαλκάνια, είναι το Συμβούλιο. Και αυτό αληθεύει ειδικά για την ΦΥΡΟΜ, διότι η Επιτροπή έχει εισηγηθεί την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εδώ και 7 χρόνια. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια ευθύνη, είναι συνυπεύθυνη κατά κάποιο τρόπο για αυτή την όθηση. Για, αυτό το αδιέξοδο, με συγχωρείτε. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να προσπαθήσετε να πετύχετε κάποια συμφωνία, κάποια ομφωνία στο Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις που έχουν αναβληθεί, να μην ε, αποτελεί ε, ξανά, να, μην υπάρχει πια αυτό το εμπόδιο. Δεύτερον, έχει αναφερθεί στην Μεσόγειο και στην Αφρική και το ε, ταμείο που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, ακολουθώ επίση την πρωτοβουλία του Ιταλού ε, Υπουργού, αλλά αυτό που έχει εισηγηθεί ήταν να συγκεντρωθούμε στο να πατάξουμε την εμπορία ανθρώπων, διότι η εμπορία ανθρώπων δυστυχώς είναι αλληλένδετη με τις μεταναστευτικές ροές των προσφύγων. Η εμπορία ανθρώπων συνεχίζεται ακόμη και στην Ευρώπη. Το τρίτο θέμα είναι το μέλλον του Βορείου Ιράκ μετά την προπτική του ISIS. Η Εσσονία θα μπορούσε να ε, ηγηθεί παρέχοντας μακροχρόνιες εγγυήσεις για το κτίσιμο της σταθερότητας σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα για τους χριστιανούς και τις θρησκευτικές μειονότητες. Ευχαριστώ τον Νικέλα, ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Θα πάω κατευθείαν στην ερώτησή μου. Θα διαβάσω μια πρόταση από αυτό το έγγραφο που τιτλοφορείται το πρόγραμμα του ε, Συμβουλίου Εξωτερικών της Εσθονικής Προεδρίας. Το τέλος αναφέρει τα εξή. Ανάλογα με την πρόοδο, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε στην ε, θητεία διαπραγματεύσεων για τον εξυγχρονισμό της Τελωνικής Ένωσης ΕΕ Τουρκίας. Νομίζω, τώρα θα μιλήσω στα ελληνικά, γι' αυτό αν θέλετε βάλτε τα ακουστικά σας. Σας δίνω το χρόνο που χρειάζεστε. Θα πω τα εξής λοιπόν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον έχουμε δύο κύριες ανησυχίες σχετικά με τον εμπόριο με την Τουρκία. Πρώτον είναι μια πολιτική ανησυχία, η δεύτερη είναι μια ε, νομική προϋπόθεση. Η νομική προϋπόθεση είναι η αναγνώριση της δημοκρατίας της Κύπρου. Ένα από τα κράτη-μέλη από την Τουρκία που βρίσκεται εκεί και χρόνια. Η πολιτική ανησυχία έχει να κάνει. Απολογούμε. Η πολιτική α, ε, ανησυχία μας είναι η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτός ο μοχλός πίεσης που έχουμε και έχει μείνει ως τελευταίος για την Τουρκία, ο οικονομικός, δεν υπάρχει άλλος, θα προχωρήσετε να τον παραχωρήσετε παραγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της Τουρκίας. Και το τελευταίο σχόλιο μου είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να μας πείτε κατά πόσον μετά την αποτυχία του ναυαγίου στην οποία, στην οποία έχετε αναφερθεί στον Κυπριακό, κατά πόσο θεωρείτε ότι η στάση που τήρησε η Τουρκία επιμένοντας σε επεμβατικό δικαίωμα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επικοδομητική στάση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Αουστρεβίτσιος. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Θα συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον Υπουργό για την Εσθονική Προεδρία με κάποια εμπειρία συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με μια προοπτική προς ε, το μέλλον. Σήμερα είναι η τελική ημέρα κύρωσης και ε, για την Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Ε, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, πήρε χρόνο, παρόλα αυτά ε, το πετύχαμε. Από την, επειδή η Σύνοδος Κορυφής θα γίνει υπό την Προεδρία σας, Τι στρατηγικό πλεονέκτημα βλέπετε στην ε, ανατολική εταιρική σχέση. Εγώ βλέπω ότι είναι μια πολύ καλή λειτουργική πλατφόρμα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας ικανοποιεί και ίσως θα μπορούσαμε να διευρύνουμε αυτή την θετική πρακτική εμπειρία από την ε, εταιρική, ε, ανατολική εταιρική σχέση με κάποιες χώρε τη Μεσογείου, της Βορείου για παράδειγμα. Θα εκτιμούσα τη σκέψη σας σε αυτό το θέμα. Και πάλι, στο θέμα των εταιρικών σχέσεων. Έχουμε σημειώσει την κοινή επιστολή της Ουκρανίας, Μολδαβίας και ε, ε, Γεωργίας ε, των Πρόεδρων των κοινοβολίων οι οποίοι ζητούν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι θέμα κινήτρων για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις κλπ. Πότε και πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ε, ε, να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υψηλές προσδοκίες. Αλλά για να προωθήσουμε το μέλλον αυτών των χωρών και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε ε, την επιτυχία τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ο κύριος πρέτα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που παρευρεθήκεστε εδώ. Έχετε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πιο νωρίς από ό,τι είχε προβλεφθεί και σε δύσκολες ε, συνθήκες όπου έχουμε διάφορες προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά κυρίως το Brexit. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις έχετε παρουσιάσει μια ρεαλιστική θέση τονίζοντας την Ένωση ε, και την ενότητα για να συνεισφέρει στην ασφάλεια των πολιτών μας. στο θέμα της μετανάστευσης και την κατοπολέμηση της τρομοκρατίας αυτό θα πρέπει να συνεχίσει με αποφασιστικότητα και αναμένουμε κάποια πρόοδα, πρόοδο στην, ε, στις συνόδους κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Αφρικής και της, ε, στρατικής, της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρώπης σε όλα αυτά τα σημεία νομίζω μπορείτε να ε, στηριχθείτε πάνω μας. Ε, τώρα, το θέμα της διεύρυνσης, ακόμη μια φορά, δεν υπάρχει αναφορά, ρητή αναφορά ε, στο, στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Έχω διαβάσει ε, αυτό που έχετε γράψει στο European West Balkans και πράγματι λέτε ότι η διεύρυνση είναι μια επένδυση, στρατηγική επένδυση για την Ευρώπη, για πρόθεση των αξιών. Θα ήταν καλό αυτό να είναι αντανακλαστικό για όλες τις ε, προεδρίες, να το αναφέρουν ρητός και να δίνουν έτσι ελπίδα και κουράγιο για την ανάληψη μεταρρυθμίσεων στις χώρες που θέλουν να ενταχθούν. Διότι εδώ και καιρό ε, μία προεδρία για ένα εξάμεινο ασχολείται με την διεύρυνση, η επόμενη ξεχνάει το θέμα. Τώρα, ως εισηγητής για τη Βοσνία θέλω να δω ε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε σχέση με την πορεία αυτής, την ευρωπαϊκή πορεία αυτής της χώρας. Πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα προετοιμάσετε τα, ε, βήματα, τα επόμενα βήματα και τι πιστεύετε σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Είναι μια, ε, μια ζωντανή συζήτηση στην ε, Βοσνία Αρζεγοβίνη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλανμόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον Υπουργό και σας εύχομαι και ό,τι καλύτερο για την ε, Προεδρία σας. Ο πρόεδρος κυβέρνησή σα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, όταν αναφέρθηκε στι προτεραιότητες τη Προεδρία, είπε ότι η Εστονική Προεδρία θα συνεισφέρει και σας παραθέτω εδώ στην προετοιμασία των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις χώρες ε, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, δηλαδή την ε, Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΑΚ Νομίζω ότι θα γίνει το φθινόπωρο στο Σαλβαδόρο, αν δεν κάνω λάθος, ε, και θα ήθελα να μου πείτε τι περιμένετε από αυτή την τόσο σημαντική σύνοδο ε, στην Αμερικανική Υπηρώ ε, τους επόμενους έξι μήνες έχετε και τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση ή τουλάχιστον τι ελπίζετε εσείς για αυτό το εξάμεινο. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια όθηση σε αυτή την ε, τόσο πολύ σημαντική διαπραγμάτευση. Άλλαξε και ο πρόεδρος στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και νομίζω ότι είναι μια ε, κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία ή την οποία τη σέρνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ολοκληρώνω στην Λατινική Αμερική υπάρχει και το θέμα τη εμβάνθησης τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μεξικού και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Χιλή. Εμεί ελπίζουμε αυτή η διαπραγμάτευση με το Μεξικό και τη Χιλή να ολοκληρωθεί εντό του εξαμήνου, δηλαδή στη διάρκεια τη Εστονικής Προεδρία. Πέραν των όσων μα είπατε λοιπόν για την γειτονία ε, στο Νότο και στην Ανατολή, θα μπορούσατε να μα πείτε και δύο λόγια για τη σχέση τη Ευρωπαϊκής Ένωση Λατινική Αμερική. Αυτέ είναι οι ερωτήσει μου λοιπόν. Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΛΑΚ Μεξικό, Μερκοσούρ και Χιλή. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, πολύ καλές ε, διεξοδικές ε, ερωτήσεις ο κύριος Λίτς τώρα. Ευχαριστώ. Σε χαρητήρια για το πρόγραμμά σας και το πλαίσιο το οποίο έχετε θέσει. Δύο ερωτήσεις σε δύο τομείς. Εδώ είμαι. Ο πρώτος τομέας είναι, εσείς ήσασταν υπουργό Άμυνα ε, στις Εστονίες και ξεκινήσατε τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Άμυνα. Υπάρχει συνεδρίαση για τον προπολογισμό και από πού θα προέρχονται τα κονδύλια αυτά. Και από ό,τι ε, φαντάζομαι πρόκειται για ένα πολύ ε, σημαντικό νέο θέμα για να ε, προωθήσετε την περαιτέρω ενότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας λέτε, αλλά υπάρχει προπολογισμό. Αν υπάρχουν θέματα προπολογισμού, το Κοινοβούλιο θα ήθελε να έχει αυτό κάποια επιρροή. Πώς βλέπετε εσείς τα θέματα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, τα εμπορικά ζητήματα και οι εξαγωγές όπλων θα πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί δεν κάνουν όλες οι χώρες εξαγωγή όπλων. Επίσης είπατε ότι θα ασχοληθείτε με τα θέματα της βιωσιμότητας. Πώς βλέπετε το πρόγραμμα ε, για τα SDGs υπήρχε ένα πρόγραμμα Εστονία 2021 για τη βιωσιμότητα. Πιστεύετε θα μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω αυτά τα θέματα, ε, διότι ε, θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίτς, ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Χρησιμοποιήστε την ευκαιρία της Προεδρίας σας για να δείξετε πόσο καλοί είστε. Ξέρω ότι είστε πολύ καλοί και καλή τύχη. Εγώ στις δραστηριότητες μου ασχολούμαι ιδιαίτερα με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και ήρθα με πολλές ερωτήσεις. Ε, αλλά μετά από αυτά που μας είπατε αυτά, ε, μου πήρατε τα λόγια από το στόμα, διότι τα είπατε όλα τόσο αναλυτικά και δεν έχω καμία επίκριση να σας κάνω. Uh, Μία συμβουλή μόνο να σας δώσω. Με βάση τα όσα είπατε, ε, η διεύρυνση ε, είναι προτεραιότητα, αλλά δεν θα κάνετε μόνο εργασίες συντήρησης, φαντάζομαι, ε, διότι η διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια γίνεται όλο ένα και πιο σημαντική για τις δραστηριότητες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επομένως θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν ε, μπορούσατε να συμπεριλάβατε και στις δηλώσεις σας και τη σημασία που προσδίδεται στη διεύρυνση. Μετά από την περιβόητη δήλωση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πριν από τρία χρόνια ότι ακόμα πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά με τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για το θέμα αυτό. Η μόνη μου ερώτηση λοιπόν είναι πώς θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Θα είναι απλώς εργασίες ρουτίνας, θα συστήσετε κάποια task force με ειδικά καθήκοντα, διότι είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε και ε, καλό θα ήταν να γίνει αισθητή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια ως ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος εταίρος. Ευχαριστώ, Ιντουαρτ Και τέλος, ε, η Ζηλάνα Ζάφκου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Όπως είπαν ήδη και οι συνάδελφοί μου, αφιερώστε μεγάλο τμήμα στη διεύρυνση και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε, αλλά ανησυχώ ε, με μία μικρή φράση που είπατε μόνο για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και είπατε ότι αυτός ο οποίος θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι οι τοπικές αρχές. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη στο γεγονός ότι ε, δεν ε, είναι μόνο θέμα διεύρυνσης και προστασίας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη σχέση με τη χώρα αυτή. Τίθεται και πολύ σοβαρό θέμα ασφάλειας. Υπάρχει μεγάλη επιρροή παραγόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Ε, σας εκλυπαρώ λοιπόν να προσέξετε πολύ περισσότερο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ε, σήμερα έχουμε και την επέτειο της Ρεμπρένιτσα. Έχουμε τη Σύνοδο στην την εφαρμογή, την αίτηση συγγνώμη της Βοσνίας Ερζεγοβίνη ε, για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουν να του δοθεί καθεστώ υποψήφια χώρα. και όπω είπε και ο κύριο Πρόντα, περιμένουμε και λύση για τον εκλογικό ε, νόμο, Αλλιώ τα πράγματα θα είναι στάσιμα στη χώρα αυτή. Σα παρακαλώ λοιπόν να την προσέξετε περισσότερο και να αναλάβετε και τα ενία ώστε να υπάρξει κάποια λύση στη χώρα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει το ηθικό πλεονέκτημα εκεί. Ευχαριστώ πολύ τη της Λένα Πριν σας δώσω τον λόγο κύριε Υπουργέ, ε, να πω και εγώ κάτι. Θα ασχοληθείτε και με την Αλβανία και τους κοσοβάρους ε, το επόμενο εξάμεινο και ε, καλό θα ήταν να θυμίζετε πάντα στους εταίρους και στους φίλους μας στην Αλβανία και στο Κωσυφοπαίδιο ότι οποιαδήποτε ε, συζήτηση για μια μεγάλη Αλβανία ε, είναι άνευ και δεν θα πρέπει ε, να ξεχάσουν τέτοιες ιδέες στα Δυτικά Βαλκάνια. Με εκπλήσει το πόσο συχνά αναφέρεται το θέμα αυτό δημοσίως και στις δύο χώρες και οι συζητήσεις για μεγαλύτερη Σερβία είναι πολύ σοβαρές και η συζήτηση για μεγάλη Αλβανία είναι ακόμα πιο ε, δύσκολη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Πολλές ε, και αφορούσαν διάφορα θέματα. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες στα 8 περίπου λεπτά. Αν δεν μπορέσω να τις απαντήσω όλες, ευχαριστώ να επανέλθω αργότερα. Ή να δώσω πιο λεπτομερείς απαντήσεις ε, γραπτός. Τέλος. Για τις ερωτήσεις ε, του κύριου Μακάνταμ για το θέμα της μετανάστευσης. Όπως είπα, μια ολιστική προσέγγιση χρειάζεται και πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση πάντα ήταν τμήμα, πώς να το πω, το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες. Πάντα υπήρχε ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που μετακινούταν είτε λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων ή για καλύτερες ευκαιρίες. Οπότε πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Εδώ πέρα συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να το πατάξουμε αυτό και ταυτόχρονα να εστιάσουμε στο πώς θα διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση και πώς θα γίνει πιο ανθρώπινη για τους ανθρώπους που μεταναστεύουν νομίμως. Αλλά Όσον αφορά τώρα τους παράγοντες που προσελκύουν τις ροές αυτές, ε, είναι περίπλοκο το ζήτημα. Και νομίζω ότι η διάσωση στην θάλασσα είναι προφανώς ε, ένα ανθρωπιστικό καθήκον ε, που προηγείται του να αντιμετωπίσουμε κάποιες αμφίβολες μήκυο που διευκολύνουν τους διακινητές να μεταφέρουν άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να έρχονται στην Ευρώπη. Είναι περίπλοκο λοιπόν το ζήτημα. Οπότε... Βεβαίω υπάρχουν ε, πράγματα ζητήματα των διασώσεων χωρίς να αποτελεί αυτό να δημιουργήσουμε έναν παράγοντα που θα προσελκύουμε ναι, και άλλους ανθρώπους. Τώρα για το μέλλον του Βορείου Ιράκ. Προφανώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Και όταν μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους ε, που επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράκ και τη Συρία, Δεν μπορούμε να θέσουμε πολιτικούς όρους, αλλά όταν μιλάμε για ανοικοδόμηση μεταπολεμική, οπωσδήποτε μπορούμε να θέσουμε όρους. Τότε θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με την ανοικοδόμηση της χώρας. Ναι, το τι θα γίνει με το μέλλον του Ιράκ ε, και της Συρίας ε, ως ε, χωρών. Πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί όταν προωθούμε την ιδέα του να επαναχαράξουμε τα σύνορα. Το μέλλον του Ιράκ και του Βόρειου Ιράκ θα πρέπει βεβαίως να εντοθεί σε σχέση με το μέλλον αυτής της χώρας και το σύνταγμα αυτής της χώρας. και βεβαίω ε, προ όφελο ε, ακριβώ των κατοίκων τη χώρα. Τώρα η ερώτηση του κυρίου Μαυρίδη για τι σχέσεις με την Τουρκία. Προφανώς η Τουρκία θα πρέπει να πληρεί τα όσα αναμένουμε από μια υποψήφια χώρα. Και οποιαδήποτε πρόοδος ε, θα πρέπει να είναι υπό τον όρο ότι θα πληρεί αυτά τα κριτήρια. Αναφέρθηκα σύντομα στην κατάσταση στην Κύπρο και στο θέμα αυτό. Ίσως ήμασταν υπερβολικά αισιόδοξοι κάποια στιγμή για τη δυνατότητα να επιληθεί το θέμα τόσο γρήγορα ε, πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Και νομίζω ότι ε, απαιτείται ε, η Τουρκία να έχει μια πιο επικοδομητική θέση για να διευκολύνει την λύση. Τώρα για το θέμα του κυρίου Αστρεβίτσιους και την Ανατολική Γειτονία νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εστιάσουμε στην εφαρμογή ε, συμφωνιών σύνδεσης ε, και ελευθεροπορίου. Μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για να προωθήσουμε το θέμα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων ε, και της ανταγωνιστικότητας και είναι επίσης και θέμα επικοινωνίας. Νομίζω ότι εστιάζουμε υπερβολικά στη συγκεκριμένη διατύπωση μεμονωμένων δηλώσεων αντί για τα πρακτικά ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών ταυτόχρονα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε χώρα έχει κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίζει τους στόχους της και να επιλέγει τον πολιτικό προσανατολισμό της και καμία τρίτη χώρα ποτέ δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις κυρίαρχες επιλογές μιας άλλης χώρας. Και η δήλωση που περιμένουμε να υιοθετηθεί στην Σύνοδο Κορφής θα πρέπει να αφορά το περιεχόμενο της ε, Σύνοδο Κορφής της Ρίχας. Λοιπόν, για το ερώτημα του κύριου Πρέντα. τον... το τι βεβαίω θα κάνουμε ως Προεδρία στις ε, διαπραγματεύσεις του Brexit είναι να ε, φέρνουμε σε επαφή τις αντιπροσωπείες του ε, κράτων μελών με τον κύριο Μπαρνιέ και να διατηρούμε την ενότητα των 27. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, τα κεκτημένα δικαιώματα των υπηκών τα σύνορα στην ίσο της Ιρλανδίας αρμοδιότητες δικαστηρίων κτλ. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να κανονίσουμε και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι μορφή θα έχει η μελλοντική σχέση, αλλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι περιορισμένος αλλά θέλουμε να διευκολύνουμε την διαδικασία. Και βεβαίω ε, δούμε και τις δημογραφικές εξελίξεις στην ε, Αφρικανική Ήπειρο. Αυτός είναι ένας παράγων ο οποίος οθεί τα άτομα Ε, μιλάμε για μια εκθετική αύξηση του πληθυσμού. Και βεβαίως ε, είναι μια πτυχή των διαφόρων κρίσεων ε, που υπάρχουν η μετανάστευση τώρα. Έχουμε ακριβώς βεβαίως και Θα ήθελα να επενέσω και τον πρόεδρο Στόντεμπελ και τις προσπάθειε που έχει κάνει και τη σκληρή δουλειά για να ξεκολλήσει η συνεργασία εκεί. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες εργασία αυτή. Ο κύριος Λίτς ε, ανέφερε ουσιαστικά το ίδιο ζήτημα και όταν μιλάμε για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο νομίζω πως ε, είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε διάφορα έργα χωρίς να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το να πάρουμε λεφτά από άλλους τομείς πολιτικής. Πρέπει να σκεφτούμε κάπως δημιουργικά. με έναν τρόπο που δεν θα εμποδίζει τους μηχανισμούς που έχουν οικοδομηθεί. Και να δούμε βεβαίω και το θέμα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας και των διαφόρων νομικών πτυχών των εξαγωγών όπλων. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις στην Προεδρία μας και παραπέρα. Τώρα, για την Σύνοδο Κορυφής, ε, η Σύνοδος ε, ΣΕΛΕΞ ε, στην, στο Ελ Σαλβαδόρ θα διοργανωθεί από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα πρέπει ακριβώς να δούμε το τι θα γίνει καθώς πηγαίνουμε προς αυτές τις Σύνοδους Κορυφής Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένες συμφωνίες στις οποίες αναφέρατε με Χιλή, Μεξικό και πάλι νομίζω πως ε, προσπαθούμε να παίξουμε έναν επικοδομητικό ρόλο για να προσπαθήσουμε ακριβώ να είμαστε επιτυχείς σε άλλα πλαίσια νομίζω θα Μπορούμε να κινηθούμε κάπως πιο γρήγορα. Το ερώτημα του κυρίου Κούκαν τώρα. Δεν θα έλεγα ότι η διεύρυνση δεν είναι πρώτη μας προτεραιότητα, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβώς ε, προσεκτικοί, ειδικά όταν μιλάμε για τις χώρες που είναι στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να δούμε ακριβώς το τι μπορεί να γίνει σε άμεσο χρόνο, αλλά θα έλεγα για Σερβία, Κοσφοπέδιο και άλλες υποψήφιε χώρες πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία όταν δηλαδή θα ανοίξει το παράθυρο ευκαιρίας ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να, είμαστε, να μας καθοδηγούν οι στρατηγικοί μας στόχοι. Και επίσης ε, να Μιλάμε πάντα με τρόπο ειλικρινή και ενώ η Ευρώπη μπορεί να μην είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για η κάποια στιγμή νομίζω θα αλλάξει αυτή η ένταξη νέων μελών, κάποια στιγμή νομίζω θα αλλάξει αυτή η δυναμική. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακριβώς και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε προς αυτόν τον στόχο. Και τέλος, ανεβοσνία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας και ότι θα πρέπει η χώρα να επιδείξει στις αρχές ακριβώς ότι υπάρχει κράτος δικαιού τώρα για προσπάθειες παρέμβαση στα ιστορικά της χώρας ε, ναι, δεν γνωρίζουμε για μένα με ενθαρρύνει κάπως ε, με κάποια πράγματα που ακούστηκαν προσφάτως αλλά Τώρα η διχαστική ρητορία όταν μιλάμε για τις ε, διάφορες ε, συνταγματικές διευθετήσεις δεν βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά οι αρχές στο εθνικό επίπεδο για να εργαστούμε επικοδομητικά Ε, νομίζω επιδεικνύουν κάποιους στόχους και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε και τέλος. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε ότι υπάρχει αυτή η ρητορία, η εμπριστική για την επαναχάραξη των συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους ε, συναδέλφους σας ε, για σε σχέση με την Αλβανία και άλλες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω ότι τα εκτιμούμε όλα αυτά. Και νομίζω ότι το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρει στην σταθερότητα στην περιοχή, μια δουλειά που οπωσδήποτε δεν έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. So good luck. Καλή επιτυχία με την Αστυνομική Προεδρία. Θα ταξιδέψετε αρκετά, θα σας δούμε στις Βρυξέλλες αρκετές φορές. Ήταν πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και Τώρα κλείνω αυτό το σημείο στην ημερήσια διαταξή μας και θα ήθελα να θυμίσω ότι το επόμενο σημείο ε, είναι και των θυρών, άρα μόνο εξοδετημένα μέλη, ε, προσωπικό των πολιτικών ομάδων και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παρευρεθούν. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους υπόλοιπους που είναι